Καλησπέρα σα αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως σα είχαμε υποσχεθεί, οργανώσαμε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Άντριου Καίτη. Ένα ε, Επίτροπος αρμόδιο για την υγεία και την επιστηστική ασφάλεια και άρα οικείο ε, στα θέματα που ενδιαφέρουν και εμάς. Σας καλωσορίζουμε εγκάρδια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την ευκαιρία αυτή που έχουμε για την ανταλλαγή απόψεων και μετά την απόφαση για τον διαρθρωτικό διάλογο με την Επιτροπή οργανώνουμε περιοδικά τέτοιες συνεδριάσεις στα πλαίσια αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου. Σήμερα έχουμε μια τέτοια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Ανδριουκάητης. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε τις ενέργειες και δραστηριότητες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και για φέτος αλλά και που προβλέπονται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017. Χαιρόμαστε για αυτή την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο και θα πρότεινα να δώσουμε πρώτα το λόγο στον αρμόδιο Επίτροπο Κάιτης για μια εισαγωγική σύντομη όχι θα το κρίνει ο Επίτροπος ομιλία μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές για τρία λεπτά στον καθένα. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο για να απαντήσει στα σχόλια των συντονιστών στις ερωτήσεις και θα ακολουθεί συζήτηση με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της συνεδρίας. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου. Σχεδόν ένα έτος έχει περάσει από τότε που ήρθα να συζητήσουμε κατά τον ετήσιο διαφρομένο διάλογο. Χαίρομαι πολύ που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω μπροστά στην Επιτροπή σας ε, σήμερα πάλι. Και σήμερα είναι πιο θετικό το πλαίσιο. Η Ευρώπη και οι γεωργοί περνούν δύσκολους καιρούς, ωστόσο παραμένω πεπισμένος ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να ενεργήσουμε από κοινού. Θα θυμάστε ότι πέρσι παρουσίασα τις προτεραιότητές μου για το σύνολο της θητείας μου. Φέτος θα ήθελα να αναφερθώ στην βιώσιμη γεωργία για υγιεινή και ποιοτική διατροφή. Πέντε θέματα θα ήθελα να αναφέρω σχετικά σύντομα για να έχουμε περισσότερο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις εκ των υστέρων. Όσον αφορά την μικροβιακή αντοχή. Κύριοι βουλευτές, γνωρίζετε ε, το πενταετές σε σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, ε, ένα πρόγραμμα που κλείνει ε, φέτος. Αυτό καλύπτεται από την προσέγγιση ενιαία υγεία. Τα αποτελέσματα τα περιμένουμε τον επόμενο μήνα, ενώ ακούσαμε και τα ενδιάμεσα, τα προσωρινά αποτελέσματα σε σχετική διάσκεψη. η νομοθετική μας πρόταση για τα κτηνιατρικά ε, φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές ε, αποτελούν σημαντικές και οικονομικέ ε, για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την έκθεσή σας για τις φαρμακούχες ζωοτροφές που παρουσιάσατε σήμερα το πρωί. Ωστόσο, απομένουν πολλά να γίνουν ε, και σας καλώ να, η Επιτροπή σας να μας στηρίξει στο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα, ε, έλεγχος κτηνιατρικών ασθενειών. Αυτό είναι σημαντικός παράγοντας για τον κτηνιατρικό και γεωργικό τομέα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις δομές και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, το θέμα αυτό και ο νέος νόμος για την υγεία των ζώων αποτελεί σημαντικό επίτευγμα στο θέμα αυτό. Τις τελευταίες δεκαετίες τα κράτη-μέλη έχουν συγκεντρώσει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών γρήπης ε, που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει προστατευτικά μέτρα για τον καθορισμό ε, περιοχών όπου επιβάλλονται περιορισμοί. Η στρατηγική καθώς και τα μέτρα για τον έλεγχο των ε, ασθενειών στόχο έχει ε, να έχουμε πληθυσμό ζώων απειλαγμένο από ιούς για την παραγωγή τροφίμων. Η βιώσιμη γεωργία σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και πιο βιώσιμο ε, τρόπο να προστατεύσουμε τα φυτά και τις καλλιέργειες μας. Ε, χρειάζονται λοιπόν οικονομικά αλλά και υγιεινά ε, ε, γεωργικά προϊόντα τα, μέγιστα, τα ανώτατα όρια καταλήπων ε, αποτελούν προτεραιότητα στο θεματολόγιο της ε, Κομισιόν και ε, τα προϊόντα φυτοπροστασίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό. Και θα πρέπει όποτε είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Σύντομα η Κομισιόν ε, θα ε, υποβάλει έκθεση με βάση τα εθνικά σχέδια ε, για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Και τέλος να αναφερθώ σε ένα επίμαχο ζήτημα, τη γλυφοσάτη. είναι ιδιαίτερα επίμαχο το αν θα πρέπει να παραμείνει στην αγορά η γλυφοσάτη ή όχι. Άκουσα προσεκτικά τις ανησυχίες, ιδιαίτερα αυτές των Ευρωβουλευτών. Έχω ακούσει πολλές ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας, την λεγόμενη έλλειψη διαφάνειας των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή οι περισσότερες ε, εκθέσεις έχουν εκπονηθεί από τον ε, σχετικό βιομηχανικό τομέα. Γνωρίζω τις ανησυχίες που εκφράζονται και για το λόγο αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την ε, από το σχετικό βιομηχανικό τομέα να δημοσιεύσει τα σχετικά του δεδομένα. Στις 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις αυτές. Να είμαι σαφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει απόφαση μόνο εφόσον υπάρχει ευρεία υποστήριξη. θα το συζητήσουμε αυτό και στη συνέχεια. Όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά πρότυπα, είναι και αυτό σημαντικό θέμα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και ιδιαίτερα ε, στη συμφωνία TTIP. Δεν παραβλέπω τις προκλήσεις, τα προβλήματα, αλλά με αισιοδοξία θα ήθελα να δω και τις ευκαιρίες που μπορεί να μας προσφέρει η συμφωνία TTIP. Ε, πρόσφατα λάβαμε πολύ ε, θετικά μαντάτα. Συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες να ξεκινήσουμε το εμπόριο δίθυρων μαλακίων. Και έχουμε πλέον τρία κράτη-μέλη που μπορούν να εξάγουν βόλιο κρέας στις Ηνωμένε Πολιτείες και επίσης προδεύουμε όσον αφορά ε, την πρόσβαση στην αγορά ε, για κάποια προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να δω όμως ίση πρόσβαση των κρατών μελών στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ενιαία οντότητα. Τέλος, όσον αφορά τις εμπορικές μας σχέσεις, να πω λίγα λόγια για την απαγόρευση ε, που έχει επιβάλει η Ρωσία για το χείριο κρέας και ε, τα σχετικά προϊόντα. Θεωρούμε ότι αυτή η απαγόρευση ε, έχει πολιτική αιτιολόγηση και καθόλου τεχνική. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη έχει αμφισβητήσει το μέτρο αυτό με προσφυγή στον ΠΟΕ. Είμαστε επεπισμένοι ότι ε, τελικά θα υπερισχύσουν τα δικά μας επιχειρήματα. Η σχετική έκθεση αναμένεται τον Ιούνιο. Ωστόσο, είμαι διατεθειμένος ε, να βρω επικοδομητική λύση και αυτό ακριβώς έχω μεταφέρει και στους Ρώσους. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι και η επόμενη γενιά θα επωφελείται από ε, υγιεινά προϊόντα διαστροφής θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, βιώσιμη γεωργία. Καταβάλουμε λοιπόν προσπάθειες ώστε να συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες στον αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής, ε, στον έλεγχο των διαφόρων ασθενειών, την ε, πιο ε, συνετή χρήση παρασιτοκτόνων και επίσης όσον αφορά την εκπόνηση των προτύπων μας, πόσο μάλλον στο πλαίσιο των, της συμφωνίας TTIP. Ξέρω ότι ε, επιγραμματικά ανέφερα κάποια θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας. Ε, θα ήθελα όμως τώρα να προχωρήσουμε στη συζήτηση και να ακούσω τις δικέ σας απόψει πάνω στα θέματα που κάλυψα και σε ενδεχομε... άλλα θέματα που θα θέλατε ενδεχομένω να θίξετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Ήταν σφαιρική η παρουσίαση των προβλημάτων. Θα περάσουμε στους συντονιστές. Τρία λεπτά ο καθένας και ξεκινούμε από τον κύριο Ντές. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή σας. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα. Όσον αφορά τα αντιβιωτικά, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την καταχώρησή τους ε, και τις διάφορες προθεσμίες. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω και στα ανθρώπινα φάρμακα να θεσπίσετε σχετικούς κανόνες. Νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στα αντιβιωτικά στον κτηνιατρικό τομέα. Ε, δεν θέλω να υποτιμήσω τη σημασία τους εκεί, αλλά ε, και στα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση ε, υπάρχει ανάγκη να παρέμβουμε. Όσον αφορά την γλυφοσάτη και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Παρακαλώ η απόφαση να ληφθεί σε επιστημονική βάση. Ε, δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις ε, με ιδεολογική βάση. Νομίζω ότι και οι μεγάλες βιομηχανίες ε, των Ηνωμένων Πολιτών δεν ενδιαφέρονται τόσο πια για αυτή την ουσία, διότι έχει λήξει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το έχουμε δει αυτό και σε άλλα προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όλα να πραγματοποιηθούν σε επιστημονική βάση. Σας ευχαριστώ και για τις εξηγήσεις σας για τη συμφωνία TTIP. Θα πρέπει να ε, φροντίσουμε να διατηρηθούν τα πρότυπά μας. Δεν φοβάμαι την TTIP, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας ε, και μας κάνατε και αυτή την παρουσίαση σήμερα το απόγευμα. Δύο ερωτήσεις ε, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτα απ' όλα τη μικροβιακή αντοχή. Είπατε ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Εμείς σε αυτή την Επιτροπή έχουμε συντάξει πολλές εκθέσεις πρωτοβουλίας και σημαντικές δραστηριότητες για το θέμα αυτό. Αναμφίβολα εξαρτάται και από την ποσότητα που δίνουμε ως τροφή στα ζώα μας, ε, κυρίως για την ε, παραγωγή πουλερικών. Δηλαδή ουσιαστικά οφείλεται στο πόσο χαμηλή είναι η ενεργειακή, η ικανότητα των τροφίμων που δίνουμε. Δηλαδή πρωτεΐνες φθηνές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα λόγω της απαγόρευσης χρήσης και για το μονογαστρικά ζώα ε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ζωικά άλευρα, είναι και θέμα ταμπού, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα και τις διάφορες προδιαγραφές ε, ναι εντάξει για τα μερικαστικά αλλά για τα μερικαστικά ε, όταν δίνουμε χαμηλής ενεργειακής περιεκτικότητας τρόφιμα δημιουργείται πρόβλημα και για τη γλυφοσάτη εάν είναι η γλυφοσάτη επιβλαβής πρέπει να σταματήσουμε τη χρήση έχει συζητηθεί πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά θέλουμε να έχουμε μια υποστήριξη από σοβαρές επιστημονικές αναλύσεις, όχι να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει εντυπώσεων ε, συναισθηματικά. Να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει επιστημονικών αναλύσεων. Οπότε εδώ ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παράσχει τέτοια επιστημονικά στοιχεία και να μας πει κατά πόσο δημιουργεί η γλυφοσάτη τα προβλήματα που αναφέρονται στον τύπο. Επ' αυτού θα θέλαμε διευκρινήσεις από εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουμε σήμερα είναι το θέμα των ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας για τα ζώα, επίσης ε, η σήμανση της χώρας προέλευσης. Μήπως ήταν καλύτερο να εφαρμόσουμε πλήρως την υφιστάμενη νομοθεσία πριν να προβούμε σε θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων. Νομίζω ότι ο πολλαπλασιασμός των νομοθετικών κανόνων δεν είναι προς όφελος κανενός, ούτε και των ε, εκτροφέων. Καλύτερα να εφαρμόζεται ομοιόμορφα η ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένης της ε, σοβούσες κρίση ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία, δεν νομίζω ότι μπορούν οι αγρότες να υποφεληθούν από νέα μέτρα όταν τα ισχύοντα δεν εφαρμόζονται ακόμη πλήρως και ομοιόμορφα. Επίσης, θα ήθελα να μα πείτε αν όλα τα κράτη-μέλη πληρούν τις προδιαγραφές για τις διαστάσεις των κλουβιών στη και το σεβασμό των διατάξεων για την ευημερία των ζώων. Επίσης, ως προς το TTIP, οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είμαστε ιδιαίτερα προσιλωμένοι στις υψηλές προδιαγραφές υγείας και ευημερία των ζώων και θέλουμε να διασφαλίσουμε αυτές τις υψηλές προδιαγραφές μας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν αντίστοιχε υψηλέ προδιαγραφέ. Οπότε πολλοί αγρότες μας φοβούνται μήπως ε, το TTIP ε, φλήση ως προς τις ε, χαμηλότερες προδιαγραφές και κατακλειστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από φθηνότερα προϊόντα που παράγονται με πιο υποβιβασμένες προδιαγραφές. Θα εξασφαλίσετε απέτηση αντίστοιχων υψηλών προδιαγραφών για τα προϊόντα κρέατος, ε, τα γαλακτοκομικά και ούτω καθεξής. Εγώ δεν πιστεύω ότι το TTIP είναι κάτι που θα δούμε βράχη πρόθεσμα δεδομένης και της πολιτικής κατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα με απασχολεί περισσότερο η κατάσταση στη Μαρκοσούρ. Ίσως αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε και να συζητήσουμε. για να μην ε, έχουμε θέμη το ανταγωνισμό ε, για τους κτηνοτρόφους μας από τους κτηνοτρόφους ε, της Μερκοσούρ, ιδιαίτερα από τη Βραζιλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι το βόλιο κρέας τη Βραζιλία παράγεται με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές, κάτι που δεν ισχύει. Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε καταράκωση της κτηνοτροφίας μας εξαιτία του ανταγωνισμού από οποιοδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Και δεν θα ήθελα να καταστραφούν οι κτηνοτρόφοι μα εξαιτία τέτοιων ατυχών εμπορικών συμφωνιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε και Χαίτεμα. Έχω τέσσερα σχόλια. Το πρώτο αφορά τα αντιβιωτικά, τη μικροβιακή αντοχή. Φυσικά χρειαζόμαστε μία πρόταση γιατί σίγουρα ε, έχουμε αυξήσει κατά 67% την κατανάλωση αντιβιωτικών. Και σίγουρα η προσέγγιση της μίας και νέας υγείας είναι πολύ σημαντική. One Health Approach. Και πολλές φορές ο κόσμος παραπληροφορείται. Νομίζει ότι ενδείκνεται για τα πάντα η χρήση αντιβιωτικών. Ακόμη και για τη γρήπη χρησιμοποιούν αντιβιωτικά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή ενημέρωση του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τα κτηνιατρικά αντιβιωτικά, αυτά που χρησιμοποιούνται για τα ζώα, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στην ευρωπαϊκή ενία αγορά ε, ομοιόμορφη ε, γιατί δεν μπορεί να έχουμε ε, ανθυγινές συνθήκες στην κτηνοτροφία και μετά να χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά για να αντισταθμίζουμε τον ανθυγινό χαρακτήρα της εκτροφής. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, 2,8 δισεκατομμύρια από την Γενική Διευθυνσάντε προβλέπονται για την επόμενη επταετία για τη χρηματοδότηση πιθανού ξεσπάσματος μιας επιζωτίας. Φαίνονται πολλά τα 2,8 δις. Αλλά αν σκεφτούμε ότι μόνο για τον αυθόδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε έξοδα ένα δις και πάνω, τα 2,8 δεν αρκούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα ασφαλίσεων κατάλληλο, γιατί αν ξεσπάσει και άλλη κρίση δεν θα έχει μείνει τίποτα στο ταμείο μας. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε ευρύτερη και ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων φυτοπροστασίας ε, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης ε, των ε, φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να έχουμε τέτοια ομοιόμορφη εφαρμογή νέων προϊόντων που επιστημονικά είναι αποδεδειγμένα ότι είναι πιο υγιεινά, έχουν χαμηλότερο κίνδυνο, θα πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερη επιλογή στους γεωργούς για να καταπολεμούν τα ζυζάνια και τα παράσιτα της αρρώσης. Έχετε μια νέα διαδικασία για τα νέα προϊόντα φυτοπροστασίας. Επίσης, υπερθεματίζω σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Δεκάστρο για την κυκλική οικονομία. Έχουμε πολλές διαθέσιμες πρωτεΐνες στο κρέας και στα κόκαλα και επίσης ε, είναι ε, υψηλής ποιότητας ε, πρωτεΐνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα πουλερικά, για τα ζώα που είναι πανφάγα και χρειάζονται και ζωικές πρωτεΐνες στο συντηρέσιο τους. Υπάρχει κάποια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε επαρκή συστήματα ελέγχου, για να μην επιτρέπονται φαινόμενα κανιβαλισμού. Αλλά δεν ξέρω, είναι δυνατόν τα πουλερικά να καταναλώνουν χειροκρές και το αντίστροφο. Γιατί έχουμε απαγορεύσει εισαγωγή σόγιας. Ε, για να μπορέσουμε να απαγορεύσουμε την εισαγωγή σόγιας. Γιατί γενετικό τροπημένη σόγια είναι πολύ χειρότερη για το περιβάλλον. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες σε εμάς πρωτεΐνες. Και άλλωστε αυτές οι πρωτεΐνες από, ε, ε, από κρέας και οστά δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνες. Γιατί λοιπόν να μην τις χρησιμοποιήσουμε. Η κυρία Σένερα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα επαναλάβω κάποιες ερωτήσεις που είχα υποβάλει και στην προηγούμενη μας συνάντηση. Από τους προλαλήσαντες ε, ε, προέκυψαν ερωτήσεις για την υγεία των ανθρώπων, για το περιβάλλον. Όταν μιλούμε για αντιβιωτικά, για παρασιτοκτόνα, για ζυζανιοκτόνα, για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να, να κυριαρχεί η αρχή της προφύλαξης. Θα πρέπει πρώτα να αποδείξουμε ότι όλα αυτά δεν είναι επιβλαβή για την υγεία. Και αυτά βρίσκονται στα χέρια της βιομηχανίας και των εργαστηρίων που χρηματοδοτούν τις έρευνες, δηλαδή Γιάννης Κερνάκη και Γιάννης Πίνη. Είναι επίγον, κατά τη γνώμη μου να έχουμε ανεξάρτητη δημόσια έρευνα που θα απαντήσει στα συγκεκριμένα αιτήματα της διαφύλαξης της υγείας και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος, της προστασίας του περιβάλλοντος. Εγώ δεν πιστεύω στην ηθική, στη δεοντολογία της βιομηχανίας και έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο κάποιες εκκρεμότητες από την προηγούμενη μας συνεδρίαση. Μία ερώτηση που δεν απαντήθηκε την προηγούμενη φορά. Ερωτώ λοιπόν, τι συμφωνίες έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την εμπορευματοποίηση μαλακίων και ποιο είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μας είπατε ότι υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά, Επίσης, ε, θυμάμαι ότι είχατε κάνει κάποιο σχόλιο στην προηγούμενη μας συνάντηση. Ρωτώ λοιπόν σε τι φάση βρίσκονται οι συμφωνίες που έγιναν σε τεχνικό επίπεδο και ποιο θα είναι και πάλι το αντάλλαγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μα ε, μας εκπλήσει λίγο το θέμα της ε, γλυφοσάτης. Ε, θα υποβάλετε νέα πρόταση διότι ακούστηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σε επιστημονική βάση, αλλά υπάρχουν δύο επιστημονικές πλευρές. Η μία που θεωρεί ότι είναι ασφαλής η γλυφοσάτη και η άλλη που δεν τη θεωρεί ασφαλή. Θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν η Κομισιόν να επιτρέψει ε, για μια δεκαπενταετία ε, την ουσία αυτή χωρίς κανένα περιορισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το θέμα, να περιμένουμε και την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Χημικές Ουσίες. Όσον αφορά τα αντιβιωτικά, αρκετοί σα ρώτησαν, θέλω και εγώ να σας ρωτήσω. Η Κομισιόν, όπω το ζήτησε και το Κοινοβούλιο, θα υποβάλει κατάλογο ε, για ε, εφεδρικά αντιβιωτικά, τα οποία δεν θα επιτρέπεται να ε, χρησιμοποιούνται στον κτηνιατρικό τομέα. Είναι επίμαχο το θέμα, θα κάνετε κάτι. Και όσον αφορά την προστασία των ζώων σε γερμανική εφημερίδα είχαμε ένα μεγάλο ρεπορτάζ για τις μεταφορές των ζώων από την Ευρώπη στην Τουρκία και ιδιαίτερα για τις συνθήκες που επικρατούν στα σύνορα της Βουλγαρίας. Αφού το γνωρίζουν και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν απαγορεύει κανείς τις μεταφορές αυτές τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι παραβιάζονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μία ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει ε, εξαγωγικές πιστώσεις σε χώρες όπως είναι η Ουκρανία για προϊόντα τα οποία ε, δεν πληρούν τα πρότυπά μας και κατόπιν επανεισάγονται προϊόντα από εκεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να υπονομεύουμε τα δικά μας συστήματα με προώθηση των εξαγωγών. Όσον αφορά την ξυλέλα φαστιτιόζα, ποια είναι η κατάσταση της καταπολέμησης. Υπάρχουν ε, βήματα προόδου ή συνεχίζει η κατάσταση να είναι εξίσου κακή. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένα. Για τη γλυφωσάτη θα ήθελα να μιλήσω αρχικά. είναι πολύ σημαντικό φυτοφαρμακό για τη γεωργία, για τη δασοκομεία και γενικότερα για διάφορες ε, δραστηριότητες, ε, ε, θα έλεγα περιφερειακές, δημοτικές. Είναι πολύ σημαντικό υλικό και αν αποφασίσετε να την απαγορεύσετε για δύο διαφορετικούς λόγους, πρέπει να δούμε και τι άλλο θα καταργήσετε. Οι λόγοι θα είναι η τοξικότητα και το ότι είναι καρκινογόνος ουσία. Τι είναι πιο τοξικό από τη γλυφοσάτη. Ξέρετε η καφεΐνη που πίνουμε είναι πολύ πιο τοξική από τη γλυφοσάτη. Το αλκοόλ που πολλοί από εμάς πίνουμε είναι πολύ πολύ πιο τοξικό από τη γλυφοσάτη. Αλλά το ρώτηνο, ε, Μαρτίν, κάτι που χρησιμοποιείται από τους βιολογικούς ε, γεωργούς είναι πολύ πιο τοξικό από τη γλυφοσάτη. Αν είναι λοιπόν να απαγορεύσετε τη γλυφοσάτη για λόγους τοξικότητας, ε, θα είμαστε, θα καταλήξουμε εμεί στη μιζέρια, διότι δεν θα μπορούμε να πιούμε καφέ, δεν θα μπορούμε να πιούμε ένα ποτό, ούτε να καλλιεργούμε βιολογικά προϊόντα. Το άλλο κριτήριο είναι ότι είναι καρκινογόνο ουσία και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είπε ότι πιθανότατα πιθανώ να είναι καρκινογόνο ουσία. Πρέπει να δούμε και τι άλλο εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Ένα από αυτά είναι το να εργάζεται κανεί σε νυχτερινέ βάρδιε. Ε, δημιουργεί καρκίνο, όπω φαίνεται. Επίσης ε, τον ε, κόβεις ε, ανθρώπινα μαλλιά είναι καρκινογόνο. Και επίσης το εθνικό πότο της Αργεντινής όπως φαίνεται. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ. Έχουμε αποφασίσει να πούμε ότι η γλυφωσάτη είναι κάτι κακό και πρέπει να το σταματήσουμε, αλλά όταν έφτασε στη, μέσα τη δεκαετία του 70, θυμάμαι ότι μας επέτρεψε, μας άνοιξε πολλούς δρόμους στη Γεωργία μας άνοιξε πολλούς δρόμους στη Γεωργία. Ε, να πω τώρα και δύο λόγια για τα ε, βιολογικά φυτοφάρμακα. Ξέρετε ότι η Αφρική μας έχει ξεπεράσει. Με δείχνετε γιατί. Δείχνετε κάποιον άλλο. Α, εντάξει. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απελευθερώσει τη χρήση των φυτοφαρμάκων ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε την Αφρική. Η Αφρική μας έχει ξεπεράσει σε αυτό σίγουρα, παρότι όχι σε άλλα πράγματα. Να αφήσετε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ε, ε, για, τα μεταλλαγμένα και ναι, τώρα για τα υπόλοιπα που είπατε για, για τα απόβλητα είναι πηγή πρωτεΐνης ε, από τα σφαγεία είναι κομμάτι της αγοράς λέτε ότι αναρωτιέμαι ποιο θα το επιλέξει, αλλά όταν μιλάμε για πηγή ε, ζωικών πρωτεϊνών, ουσιαστικά ε, τα έντομα δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κανονισμό για τα σφαγεία. Μάρτιν, ε, σας υποστηρίζω για αυτό το ζήτημα της μεταφοράς των ζών των ζώων. Είναι αποκρουστικό αυτό που συμβαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ντρέπεται για ορισμένες από που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρο. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο των σχολείων από τους συντονιστές. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο για να απαντήσει και θα ακολουθήσει γύρος ερωτήσεων με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πολλοί συντονιστές ε, έθεσαν παρόμοια ερωτήματα. Τη γλυφοσάτη, τη μικροβιακή αντοχή, το TTIP συνέπεσαν ε, γενικώ ερωτήσεις και υπέβαλα και πιο ειδικέ μερικές φορές παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά την μικροβιακή αντοχή στα αντιβιωτικά. Όπως ξέρετε, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ και των δύο πλευρών, και της κτήνετρικης ε, πλευράς και της πλευράς της ανθρώπινης υγείας, και της υγείας των ζώων και της υγείας των ανθρώπων. Επίσης, να δούμε και το περιβαλλοντικό σκέλος. Υπάρχουν πολλές συνιστώσεις εδώ στο πολυδιάστατο αυτό ζήτημα της υγείας. Αναφέρατε ότι γίνεται κατάχρηση ή υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών από ανθρώπους. Και όντως σε μερικές χώρες έχουμε είτε κατάχρηση είτε υπερβολική χρήση αντιβιωτικών για προβλήματα ανθρώπινης υγείας. Έχουμε όμως μερικές φορές καταμένη χρήση αντιβιωτικών και στην κτηνοτροφία. Εγώ θα ήθελα να δημιουργήσω μια πλατφόρμα ενιαίας υγείας, της μίας και μοναδικής υγείας, με συμμετέχοντες από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Και μάλιστα ε, σε μια Ολλανδική διάσκεψη συμμετείχαν και Υπουργοί Υγείας και Υπουργοί Γεωργίας και ήταν πολύ καλό αυτό το παράδειγμα και πρωτοφανές και υπόδειγμα για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υγεία ως ενιαίο φαινόμενο σε όλους τις πολιτικές και να συσπηρωθούμε να ε, μαζέψουμε τις δυνάμεις μας και φυσικά να ακολουθήσουμε τους επιστήμονες και τα επιστημονικά πορίσματα. Ο κύριος ΔΕΣ μίλησε για μια προσέγγιση που θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά πορίσματα. Εννοείται. Και φυσικά ε, χρειαζόμαστε και μια νέα μεθοδολογία για να ε, χαρακτηρίσουμε τη χρήση, την κατάχρηση, την υπερβολική χρήση και επίσης ε, ε, κοινά συστήματα παρακολούθησης, ε, ιχνηλασιμότητας και να βελτιώσουμε και τις νομοθετικές μας διατάξεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα, τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα θέματα για την ανθρώπινη υγεία. Και να μην ξεχνούμε ότι εκπνέει στα τέλη του 2016 και το σχέδιο δράσης για τη μικροβιακή αντοχή. Οπότε θα πρέπει να ανανεωθεί. Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Ιούνιο για το τι μέλη γενέστε και ποιος θα είναι ο ακολουθητέος δρόμος. Πάντως θα πρέπει να έχουμε και τα συμπεράσματα των δύο συμβουλίων υγείας και γεωργίας. Πάντως αυτή είναι η καλή ευκαιρία για να αναδειχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, καλύτερο τόπο για βελτίωση του ελέγχου σε ό,τι αφορά τη χρήση των αντιβιωτικών και στους ανθρώπους και στα ζώα. Επίσης, ε, τα περιβαλλοντικά θέματα. Ξέρουμε εκεί που παρασκευάζονται οι φαρμακούχες ε, ζωοτροφές ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εκεί. Τι μεθοδολογία χρησιμοποιείται και πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε και τις επιρροές στο περιβάλλον. Και σε τρίτες χώρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Και στις ε, συζητήσεις που έχουμε διεθνώς θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των εταίρων μας και στο θέμα αυτό. Είχα πάει στην Κίνα και είχα επισημάνει αυτά τα θέματα σε συναντήσεις που είχαμε τις Κινέζικες Αρχές. Το ίδιο και σε συναντήσεις που είχαμε υπουργού από τη Βραζιλία, από τις Ηνωμένε Πολιτείε και εκεί επισήμανα αυτά τα θέματα. Και θα το συζητήσουμε και στο TTIP για να ενθαρρύνουμε και τις άλλες χώρες εταίρους να δραστηριοποιηθούν για την πάταξη της μικροβιακής αντοχής. Θα πρέπει να δείξουμε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ενεργές και δραστήριες ό,τι αφορά την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Πάντως θα συνεχιστούμε με παραλίλου συζητήσεις για τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και θα προωθήσουμε καλύτερο διακλαδικό διατομιακό διάλογο στα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να, συζητήσουμε, να και ένα δίκτυο μικροβιακής αντοχής μεταξύ των κρατών μελών για να προωθήσουμε έρευνα και καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη για την αναζήτηση και παρασκευή νέων φαρμάκων και να προωθήσουμε γενικώ τις προσπάθειες. Αυτά για την μικροβιακή αντοχή, το AMR. Τώρα, για το TTIP. Επιβεβαιώνω ότι συνεχίζονται καλά οι διαπραγματεύσεις για το φυτογειονομικό και υγειονομικό σκέλος. Φυσικά, θα πρέπει να προσπίσουμε τις προδιαγραφές μας και μέσω του TTIP θα έχουμε ευκαιρίες για καλύτερες εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε θέματα γεωργίας και γεωργοεπιστηστικά. Το TTIP όμως δεν αφορά μόνο ε, προδιαγραφές ασφάλειας ε, τροφίμων. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της συζήτησης του TTIP, οι προδιαγραφές της ασφάλειας των τροφίμων. Είναι σαφές σαφέστατο ότι θα πρέπει να προασπίσουμε, να διαφυλάξουμε τις προδιαγραφές μας για την ασφάλεια τροφίμων, τους νομοθετικούς μας μηχανισμούς, του, τους ελεγκτικούς μας μηχανισμούς, τους μηχανισμούς αξιολόγησης και να πρόκειται σε εμά να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τις Ηνωμένε Πολιτείε στα Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το πιο δύσκολο θέμα είναι να ενθαρρύνουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε να δεχθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία και ενιαία οντότητα. Γιατί τα υγειονομικά και το φυτοϊγειονομικά μέτρα, να τα σκεφτούμε ως μέτρο, ως τρόπο για να το προωθήσουμε αυτό είναι δύσκολο, γιατί υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξάγουν τα αγαθά τους προς τις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 28 χώρες μέλη και δεν έχουν καμία δυνατότητα να είναι σε ίδια θέση. Από εμά τώρα, αν ξεχωριστά οι χώρες εξάγουν ε, βόηο, κρέας, ε, μερικές έχουν τέτοιο δικαίωμα και άλλες όχι. Υπάρχει μεγάλη συμμετρία και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για μας. Τώρα, για συγκεκριμένες ερωτήσεις ως προς την ως τύπη, γαλακτοκομικά προϊόντα ή μαλάκια. Μετά από μια ε, μεγάλη διαδικασία ελέγχου το, της ισοδυναμίας, έχουμε το σύστημα για την παραγωγή μαλακίων ή ισοδύναμων μεθόδων επισητιστικής ασφάλειας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και συμφωνήσαμε και οι δύο πλευρές ε, ότι έχουμε ισοδύναμα συστήματα. Και το αποτέλεσμα το αίσιο θα ήταν να βρούμε αμοιβαία ισοδυναμία. Εμείς είπαμε ότι μόνο με ισοδυναμία θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τις πόρτες και από τις δύο πλευρές για ε, εισαγωγές και εξαγωγές ε, οστρακοειδών και μαλακίων. Τώρα όσον αφορά το γάλα, όπως ξέρετε, σήμερα τρία πιλωτικά κράτη-μέλη, η Κατοχώρηση Γαλλία και η Ιρλανδία, ελέγχθηκαν από ε, τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμακών των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών μας έχουν ρωτή, ε, τους έχουμε ρωτήσει για την πρόοδο αυτού του φακέλου και γνωρίζουν το πόσο ενδιαφέρονται ε, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό έχει αναφερθεί σε συζητήσεις ε, γεργικού θέματος ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συζήτησα εγώ όταν το Δεκέμβριο του 2015 επισκέφθηκα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αναμένουμε από πλευράς τους να μας πούν τα σχόλιά τους. Αλλά η αμοιβαία ισοδυναμία αποτελεί βασική αρχή και για τις δύο πλευρές ε, ε, κανονιστικά ζητήματα. Ε, κάποια ερωτήματα ακούστηκαν σε σχέση με την ε, ξυλέλα Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ε, έχω συναντήσεις ε, με ε, τον Ιταλό Υπουργό, τον Γάλλο Υπουργό για να παρακολουθούμε την ε, κατάσταση και για να συζητάμε το τι πορεία θα ακολουθήσουμε, διότι από την Ιταλική πλευρά ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με μια απόφαση του δικαστηρίου στην περιοχή της ε, Πούλια και σταμάτησαν την εισαγωγή ορισμένων απαραίτητων μέτρων. Αλλά αναμένουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου σε μερικούς μήνες. Ωστόσο προς το παρόν πρέπει να γίνει επιτήρηση της περιοχής από την πλευρά μας. Το 2015 διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει πλέον ε, κανένα άλλο έβρεμα εκτός από ένα στην Πούλια στην Ιταλία και ένα στην Κορσική και στην περιοχή της Προβυγγίας Άλπαιων ε, στη Γαλλία η Επιτροπή προσαρμόζει τα μέτρα της ώστε να είναι βέβαια ότι είναι πάντα αναλογικά λαμβάνοντας ε, την εξέλιξη των κρουσμα... υπόψη την εξέλιξη των κρουσμάτων με σκοπό την εκρίζωση του βακτηρίου ή την αναχέτηση της εξάπλωσής του προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είχα την ιδέα να διοργανωθεί μια συνάντηση υψηλού επίπεδου όπου θα προσκαλέσουμε υπουργού ε, των μεσογειακών χωρών Ελλάδας, Μάλτας, Κύπρου, Κροατίας, Σλοβενίας, Γαλλία, Ισπανίας και Ιταλίας ώστε να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά, το πώς θα διαχειριστούμε σωστά το κρούσμα του βακτηρίου ξυλάλα αλλά θα πρέπει να αναμένουμε και την τελική αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διότι θα αποτελέσει σημαντικό γεγονός το να δούμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Κάποιοι έκαναν ερωτήσεις σε σχέση με τη γλυφοσάτη. Θα ήθελα να πω Ναι, κύριε, ο κύριος Χόισλινγκ ανέφερε δύο οργανισμούς, ΕΦΣΑ και ΑΙΑΡΚ. αλλά πρέπει να πω ότι σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ε, έχουν φτιάξει μια επιτροπή παρακολούθησης των φυτοφαρμάκων και αυτοί αξιολογούν τις επιπτώσεις της γλυφοσάτης και είχαν άλλη γνωμοδότηση σε σχέση με την ΕΑΡΚ ε, και πιο κοντινή στην ΕΦΣΑ. Επτά διαφορετικοί, δηλαδή οργανισμοί εθνικοί, είχαν επτά διαφορετικές προσεγγίσεις και και έχουν την άψη ότι η γλυφοσάτη ίσως να είναι πιθανός ε, καρκινογόνος αλλά πολλοί οργανισμοί αξιολόγηση είχαν διαφορετικές απόψεις και όχι μόνο υπό την επίρρεια της βιομηχανίας όπως πολύ συχνά αρεσκόμαστε να λέγουμε αλλά όσον αφορά την ευαισθησία του θέματος και τη σημερινή κατάσταση και τις σχετικές δυσκολίες πρέπει να πω ότι είμαι έτοιμος να αξιολογήσουμε την κατάσταση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το σύστημα αξιολόγησής μας ώστε να το καταστήσουμε πιο διαφανές δημοσιοποιώντας αυτές τις μελέτες της βιομηχανίας γιατί χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Χρειάζεται να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη. Διαφορετικά είναι δύσκολο να διαχειριστούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την κατάσταση ακολουθώντας αυστηρά και μόνο ε, επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή συζητάμε το ζήτημα ως κράτη-μέλη. Στη μόνιμη επιτροπή, ξέρετε, ακούστηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις ε, από το κάθε κράτος μέλος. και εμείς δεν διατηθέμεθα να προχωρήσουμε χωρίς απόψεις των κρατών μελών, χωρίς την ε, συγκατάθεσή τους. Πρέπει να υπάρχει κοινή ευθύνη. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε. Θέλουμε μια σαφή κατανοητή θέση και από τα 28 κράτη-μέλη. Θέλουμε μια ευρεία συμμαχία για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση για τη Λιφωσάτη. Επίσης, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, η ΕΦΣΑ παρουσίασε κάποιες απόψεις ότι κάποιοι τύποι είναι, κάποιες, συνθε... Ε, ε, ε, ενώσεις είναι πολύ επικίνδυνες και πρόκειται να προτείνει την απαγόρευση κάποιων ενώσεων αλλά σε διάφορους βαθμούς ευελιξίας ανάλογα με θέματα βιοπικιλότητας το ενδεχόμενο μείωσης του χρόνου ε, παράτασης, ε, της παρακολούθησης, διαφορετικές προσεγγίσεις. Ε, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι μια κοινή θέση των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνη τη. Δεν είναι σωστό η διαδικασία αυτή. Οπότε φυσικά το, Ευρωπα... το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γλυφοσάτη επίσης είναι σημαντικό. Ήθελα να τα αναφέρω αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε αυστηρά επιστημονική προσέγγιση. Αναφέρθηκαν και τα ζητήματα των ζωικών πρωτεϊνών. Ναι, το κοινό ερευνητικό κέντρο εξετάζει το κείμενο και θα αναλύσουμε την έκθεση και θα δούμε τι απόφαση θα λάβουμε. Επίσης ανέφεραν ορισμένοι κάποια θέματα που σχετίζονται με τις ε, ζωονόσους ε, ζητήματα δημοσιονομικά. Ξέρετε κάτι, συγγνώμη, αλλά εσείς τα είπατε τα νούμερα αυτά, δεν είναι αλήθεια 2,8 δισεκατομμύρια, μόνο 140 εκατομμύρια ευρώ έχουμε για την επταετή περίοδο. Δηλαδή 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό για τα τρέχοντα φυτογεωνομικά μέτρα. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα ε, να ζητηθούν και τα ζητήματα διασφάλισης, αυτά συζητήθηκαν και τα αποτέλεσματα ήταν αρνητικά είναι πολύ δύσκολο να εισαχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πολύ δύσκολο στη διαχείριση και ούτω καθεξής. Πολύ δύσκολο να δι... εφαρμοστεί όπως το έχουμε σήμερα. Τώρα γενικότερα για την καρυλή μεταχείριση των ζώων, η θέση μας, και εσείς αναφέρετε και τις εξαγωγές των ζώων μας σε ορισμένες χώρες και τα σχετικά προβλήματα, όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και τα σχετικά πρότυπα. Ξέρετε, τα πρότυπα αυτά έχουν συμφωνηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων και στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Εμείς επικοινωνούμε με τρίτες χώρες, είμαστε διατεθειμένοι για τέτοια επικοινωνία. Για τα ζητήματα του βόηου κρέατος ε, στη Βραζιλία, για παράδειγμα, Ξέρετε ότι είμαστε διατεθειμένοι να στείλουμε ελεγκτές σε τρίτες χώρες αυτή για να δούμε, να διαπιστώσουμε κατά πόσο ε, ε τηρούν τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και όποτε συζητάμε ε, οτιδήποτε με τρίτες χώρες πάντα θίγουμε το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων και τα σχετικά πρότυπα αλλά φυσικά δεν μπορούμε εμείς να απαγορεύσουμε την εξαγωγή σε τρίτες χώρες όπως προτάθηκε εδώ διότι είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή μια τέτοιας απαγόρευσης υπό τέτοιε συνθήκες. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε 20 ε, συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Προτείνω ένα λεπτό στον καθένα. Και να καλωσορίσω και τους επισκέπτες του κύριου Νταντά από τη Ιαπωνική Σχολή του Σαμπέρι. Καλώς ήρθατε και χαιρόμαστε που μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Ο λόγος στην κυρία Νταμάτο πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω ε, για κα, κάποιες διευκρινήσεις. Ε, θέλω δηλαδή πιο, πιο από τον Επίτροπο, αν είναι δυνατόν, δεδομένης της απόφασης του δικαστηρίου που εκκρεμεί επί της νομιμότητας των μέτρων αντιμετώπισης της ξυλέλα στην Πούλια και πάρα πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο το βακτήριο είναι καρκινογενές για τα ε, ελαιόδεντρα αποφασίστηκε να εφαρμοστούν οι αρχές της ε, λογικής και της ε, αναλογικότητας σύμφωνα με την οδηγία 29.000 τι θα κάνει με τη διαδικασία επί δηλαδή της Ιταλίας η Κομισιόν δεύτερη ερώτηση για τη γλυφοσάτη Απαντήσατε εν μέρη. Είπατε ότι θα ζητήσετε από τη βιομηχανία να δημοσίευσει πληροφορίες ε, σε σχέση με τι μελέτες. Κάντε κάτι παραπάνω. Χρησιμοποιήστε το κανονισμό 1107 του 2009 και ζητήστε δυνάμει αυτού για το δημόσιο συμφέρον να επιβληθεί στην ΕΦΣΑ η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών πριν ε, οποιαδήποτε άλλη ανανέωση, ακόμη και αν είναι μόνο για 8-10 χρόνια, ε, γίνει οποιαδήποτε άλλη ανανέωση της άδειας κρίσης της λιφωσάτης για άλλα 8-10 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε και στην οθόνη πίσω και μπροστά σας στη μικρή οθόνη το χρονόμετρο και παρακαλώ μην υπερβείτε το λεπτό καθένας. Ο κύριος Έρντος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σκάνδαλο παρόμοιο με αυτό του αλογίσιου κρέατος. Χθες συζητήσαμε το θέμα αυτό. Η 29% του μελιού που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νοθευμένο και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες επισήμανσης, διότι αυτή τη στιγμή η ετικέτα πρέπει να γράφει εάν το μέλι προέρχεται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες ή αν είναι μείγμα μελιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τρίτες χώρες. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους συναδέφους να υποστηρίξουν την ιδέα, το Ευρωκοινοβούλιο, να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Στην παρουσία σας ε, αναφερθήκατε στην πρόληψη. Θα ήθελα στο όνομα των Ολλανδών ε, εκτινοτρόφων. Ε, θα ήθελα να ακούσω τι κάνετε για τον πολύ μεγάλο αριθμό καρκίνων στην Ευρώπη και θα πρέπει να παραταθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η πρόταση του 2005 για τον ε, αμίαντο. Και επίσης είσαστε διατεθειμένοι να προσφέρετε επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στα, ε, στις γεωργικές περιοχές. θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τις συνδυάσουμε με την αποτελεσματική αφαίρεση του αμίαντου. Ε, μιλήσατε για πρόληψη, ελπίζω όμως να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που μας δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και υποβολή ερωτήσεων. Και ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχετε με την Επιτροπή μας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικώ. Έχω πολλές ερωτήσεις. Η Πολωνία, η Λιθουανία και οι Βαλτικές χώρες γενικώ επηρεάστηκαν και επλήγησαν από την πανόλη των χείρων. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Υπέθρου μας ρωτάνε πότε επιτέλους αλλάξει η κατάσταση. γιατί έχουν επηρεαστεί πολλά κοπάδια χείρων από την Αφρικανική Πανόλη των χείρων και ο κόσμος, οι κτηνοτρόφοι, οι χειροτρόφοι φοβούνται. Ε, γιατί αυτό επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος και δεν θα έχουμε ποιοτική κτηνοτροφία και υψηλές προδιαγραφές αν δεν έχουμε αρκετούς πόρους. Και μάλιστα στείλαμε και επιτροπή στον πρόεδρο Γιουνκέρ επισημένοντα τα προβλήματα των χειροτρόφων ειδικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να του βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, όσον αφορά τη γλυφωσάτη θα ήθελα η απόφαση να ληφθεί με επιστημονική βάση. Πιστεύω ότι τουλάχιστον ε, τα κράτη-μέλη ε, να πούνε ποια είναι η θέση τους και όχι με αποχή να αναβάλουν την απόφαση. Όσον αφορά το εμπάρκο της Ρωσίας, ε, χαίρομαι που είπατε ότι σας ενδιαφέρει και σας μια επικοδομητική λύση. Είναι σημαντικό να εξαλείψουμε τα εμπόδια αυτά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εργαστούμε επικοδομητικά και για να λύσουμε το πρόβλημα των μαύρων ληστών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντριέ, ευχαριστώ και ευχαριστούμε και τον Επίτροπο που ήρθε. Η γεωργία και κυρίως η αμπελουργία και η παραγωγή απορροκυπευτικών παραπονιούνται για την έλλειψη εναρμόνισης της νομοθεσίας ό,τι αφορά την εμπορευματοποίηση φυτογενομικών προϊόντων, κάτι που στρεβλώνει τον εσωτερικό ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες ζώνες. Ξέρω ότι σας απασχολεί το πρόβλημα και διερωτώ με αν θα προτείνετε μέτρα για την αντιμετώπιση του. Αναφερθήκατε και στον έλεγχο των επιζωτιών. Είπατε ότι θέλετε να βοηθήσετε τους μηχανισμούς για τον έλεγχό τους. Ε, θυμάστε τη γρήπη των πουλερικών στην Ανατολική Γαλλία και είχαμε κινητοποίηση του ε, Υπουργείου. Ήταν, σημαντική, ήταν σημαντικός ο περιορισμός τοπικός για να μην ε, έχουμε διάδοση της επιζώτιας. Χρειαζόμαστε όμως μηχανισμούς και εργαλεία. Αλλά καλό θα ήταν να έχουμε εργαλεία που να αντιμετωπίζουν και την αιστεία για τα πτηνά ε, και ιδιαίτερα τα υποαστήρια και τους εκτροφείς και να έχουμε έναν σημαντικό κοινοτικό μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε τον οικονομικό και, ε, ε, τον ε, οικονομικό και τον υγειονομικό αντίκτυπο και να αντιμετωπίζουμε τέτοιες κρίσεις. Η κυρία Νόιχρου. Σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, ε, σας ενδιαφέρουν ε, τα πρότυπα για την υγεία ανθρώπων και ζώων και για την προστασία των ζώων. Ε, αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των των καταναλωτών και των ζώων. Γι' αυτό στο θέμα της γλυφοζάτης θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης. Και όσον αφορά την χρήση αίματος αλόγων, ξέρετε ότι σε μεγάλο βαθμό εισάγεται το αίμα αυτό το οποίο χρησιμοποιείται στην χειροτροφία, το οποίο όμως ε, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Ε, θα ε, ήθελα επιτέλους στον τομέα αυτόν να αναλάβουμε, ενέργεια, να αναλάβουμε δράση ώστε να ελέγχεται το αίμα εξίσου με το κρέας. Και επίσης θα ήθελα να μου απαντήσετε όσον αφορά τον ευνουχισμό των ε, χείρων χωρίς ε, αναισθητοποίηση, τι γίνεται, υπάρχει κάποιο πρακτικό σχέδιο, δεν με ενδιαφέρουν απλά οι συλλογισμοί σας για το θέμα, με ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί έχουμε και το σφυράκι του Πρόεδρου που με τρομάζει λίγο. Η μικροβιακή αντοχή ξέφυγε ένα πράγμα. Ξέχασα μια ερώτηση ενό προηγούμενου συναδέλφου επίτροπο Θα προβλέψετε κάποιο κατάλογο των αντιβιωτικών που θα προορίζονται αποκλειστικά για την ε, ε, ανθρώπινη διατροφή, για τους ανθρώπους. Όσον αφορά τη γλυσοφάτη, πολλέ φορέ έχουμε αναφερθεί, και το είπατε κι ε, στην αναγκαιότητα συμφωνία με το Συμβούλιο, αλλά πολλά κράτη-μέλη όπω η Ιταλία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Ολλανδία έχουν δώσει αρνητική γνώμη. Δεν θα έπρεπε να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης αφού υπάρχει και επιστημονική βάση, επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ε, ε, την ακαταλληλότητα αυτού του προϊόντος. Τέλος για την ξυλέλα. Όπως είπαμε, υπάρχει, ε, δεν, δεν είμαστε επιστημονικά βέβαιοι για την ξυλέλα και τις επιπτώσεις της. Εσείς μας διαβεβαιώσατε ότι δεν έχουν ε, εντοπιστεί νέα κρούσματα. Μήπως θα ήταν καλό επειδή η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται πάλι, μήπως θα ήταν καλό να αρχίσουμε να επιτρέπουμε την φύτευση νέων ελαιόδενδρων στις ε, ζώνες που επλήγησαν περισσότερο. Ευχαριστώ. κυρία Μίλλερ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ μιλήσατε για περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας. Νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η γεωργία και ε, μας προμηθεύει με ε, υψηλής ε, αξίας προϊόντα τα τρόφιμα μας ενδιαφέρουν κυρίως. Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, να ρωτήσω τι γίνεται με τα εισαγόμενα ζώα και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως προβλέπει μέτρα για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων Επίσης, ε, όσον αφορά την γρήπη των πουλερικών και ε, την γρήπη των χείρων, με ενδιαφέρει επίσης να ασχοληθούμε με την φυματίωση. Όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή, θα ήθελα να σας πω ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε και με ε, τα υγρά ανθρώπινα απόβλητα, διότι και στα νοσοκομεία για παράδειγμα, διότι δεν ε, υπάρχουν εγκαταστάσεις ούτε στα νοσοκομεία επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ε, τα οποία όμως ε, περιέχουν πολλά μικρόβια, ορμόνες κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεμπαστιά. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, πέρυσι εντοπίστηκαν πάρα από 100 κρούσματα ενός παρασίτου στα εσπεριδοειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μαύρων κοιλίδων. Οι περισσότερες ε, ε, ήταν από την Αφρική. Και πέντε κρούσματα να εντοπίσουμε πρέπει να αναλάβουμε αμέσως μέτρα. Ξέρετε ότι αν περάσει αυτή, αυτό το παράσιτο στην Ευρώπη από την Αφρική θα μείνουν στήρα τα δέντρα και θα καταστραφούν οι παραγωγές περιδοειδών. Θα αναλάβετε επιτέλους δράση για το black spot των εσπεριδοειδών. Επίσης, οι νέες, οι νέοι, οι μέθοδοι βελτίωσης των φυτών προβλέπουν γενετική τροποποίηση. Ε, προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση αυτών των νέων τεχνικών βελτίωσης, ώστε να ε, συμπεριληφθούν στην νομοθεσία των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Θα ήθελα μία σαφή απάντηση γι' αυτό, για τις νέες μεθόδους βελτίωσης. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια απέρριψε την πρόταση ε, του κανονισμού το 1829 ε, για τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς ε, στα τρόφιμα ή στις ζωοτροφές. Δεν μείναμε ικανοποιημένοι από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών είναι ιδιαίτερα προβληματικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ επίμαχο και δεν υπάρχει ενιαία θέση αλλά διάσταση απόψεων. Ε, έμειναν ε, δυσαρεστημένοι και αυτοί που είναι κατά των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, αλλά και οι υπέρμαχοι. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επέτρεψε τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις για την απαγόρευση ή για τον περιορισμό εισαγωγής γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Επίσης, η πρόταση αυτή δεν έλυσε σωστά το θέμα της παραβίασης ε, του, της ενιαίας αγοράς με την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από τρίτες χώρες. Πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νέα πρόταση σχετικά και αν ναι, πότε. Επίσης, ε, μια και 150 περιοχές και 4.500 ε, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει ότι είναι απαλλαγμένοι από γενετικός τροποποιημένους οργανισμούς. Διαρωτώμε πώς θα, πότε θα δώσετε επιτέλους την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν κυρίαρχα και αυτόνομα αποφάσεις για τα θέματα των γενετικών τροποποιημένων οργανισμών χωρίς περιορισμούς ε, ή οποιαδήποτε εμπόδια. Η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος ε, δεν καταφέρει να συμμετάσχει στο σεμινάριο για την ευημερία των ζώων σήμερα το πρωί και αυτό είναι κρίμα γιατί αν είχε συμμετάσχει θα είχε ακούσει τους υπουργούς του Βελγίου, της Γερμανίας, της Δανίας, των, ε, της Σουηδίας, ε, των κατοχωρών που θέλουν αυστηρά μέτρα για την προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων, για να υπάρξει μια πραγματική στρατηγική σε θέματα προστασίας της καλής μεταχείρισης των ζώων. Και όλα αυτά εντός ενός νόμου πλαισίου αυτό ξεπερνά τα όσα μας προτείνει η Sanko και η Επιτροπή ε, οι οποίοι περιορίζονται με κάποιες επαφές με τους ενδιαφερομένους, κάποιους ελέγχους, κάποιες πλατφόρμες. Ε, δεν είναι αρκετά όλα αυτά. Πώς λοιπόν πρόκειται η Κομισιόν να ανταποκριθεί στις επιθυμίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να έχουμε μια πραγματική στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων και αφού έχω το μικρόφωνο για να κλείσω, πριν κλείσω, μια ερώτηση για την νομιμότητα του ανταγωνισμού. Πολλοί συναδελφοί λένε ότι η εισαγωγή προϊόντων ε, ε δεν υπάρχει, εισάγονται προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στους, ε, στα πρότυπα. Λέτε εσείς ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρξει υποβαθμίση προτύπων, αλλά πώς θα το κάνετε όλο αυτό. Εμείς με τις επιχορηγήσεις προωθούμε και ενθαρρύνουμε τις εξαγωγές, ε, για παράδειγμα, προϊόντων ε, που επανισάγουμε μετά πώς μπορείτε να δέχεστε να εξάγουμε τέτοια προϊόντα και μετά να τα επανεισάγουμε. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τον Επίτροπο. Γιατί μια τόσο απλή διαδικασία όπως είναι η αμοιβαία αναγνώριση δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Γιατί κάτι που ενώ θεωρούμε ότι είναι τόσο απλό δεν λειτουργεί, μία αναγνώριση των φυτογεωνομικών προϊόντων ε, στις ε, συναλλαγές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Τι μέτρα πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχανισμό με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί να έχουν τα ίδια μέσα ε, και προϊόντα για να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους σε ό,τι αφορά τους ενδοκρινολογικούς ή ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πώς έχει ή ενδοκρινικους διαταράκτες. Πώς έχει κατάσταση, κύριε Επίτροπε, συγκεκριμένα, τι γίνεται με τη μελέτη επιπτώσεων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η μελέτη. Και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το σωστό και σαφή συγκεκριμένο ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Επίσης, συμφωνώ και ε, εστερνίζομαι την ε, ερώτηση του κυρίου Σεμπαστιά. Φαίνεται ότι εισάγουμε από την Νότια Αφρική το παράσιτο black spot ε, που προκαλεί τεράστια προβλήματα στις περιδοειδείς, στις καλλιέργειες περιδοειδών. Θα λάβετε μέτρα κατά των εισαγωγών από την Νότια Αφρική προκειμένου να μην επεκταθεί αυτό το παράσιτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γεωργία είναι πολύ άριθμα και για να επιληθούν ορισμένα από αυτά θα απαιτηθούν ε, οικονομικές προσπάθειες από συμβουλή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά για την αντιμετώπιση άλλων χρειάζεται να υπερβούμε διοικητικά ε, εμπόδια. Ε, το χείριο κρέα στη Ρουμανία έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο λόγω του ρωσικού εμπάργου, αλλά και λόγω του ε, εμπορίου ζών χειρών εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αυτό είναι δυνατό με τρίτε χώρε από το 2013, είναι αδύνατο εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι το 2007 στη Ρουμανία εντοπίσαμε ε, περιπτώσεις Πανόλη των χείρων αλλά οι αρχέ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίζεται η υγεία των ζώων και η ασφαλεία των τροφίμων. Ξέρω ότι κάνατε μια συζήτηση τον Ιανουάριο με το Υπουργείο Γεωργίας και είπατε ότι θα ξεμπλοκάρετε ε, θα απελευθερώσετε, θα ανοίξετε αυτό το εμπόριο των ζώων των χείρων. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Σύντομη ερώτηση. Πώς θα εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τα φυτογειονομικά επιτρέπει την απαγόρευση ενός προϊόντος σε μια χώρα λόγω του κινδύνου, αλλά στη διπλανή χώρα επιτρέπεται ακόμη και στη βιολογική γεωργία. Ευχαριστώ κυρία Μόη. Η κυρία Μόη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα να αναφερθώ στη Λιφωσάτη και να σας ρωτήσω ε, να μας πείτε εκ μέρους της DJ Agri είναι δυνατόν πριν η Κομισιόν λάβει την τελική απόφαση ή ολοκληρώσει το σχέδιο, είναι δυνατόν να διεξαχθεί μια σοβαρή επιστημονική μελέτη, γιατί εσείς προηγουμένω είπατε ότι για το θέμα αυτό της γλυφωσάτης και των ενδεχόμενων αδειοδοτήσεων για το μέλλον χρειάζονται επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να λάβουμε αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Διότι από όσο ξέρω εγώ, η άποψη της ΕΦΣΑ στην οποία βασίστηκε η Κομισιόν για το σχέδιο της βασίστηκε σε έξι μελέτες που χρηματοδότησαν εταιρείε οι οποίες ούτως ή άλλως εμπορεύονται αυτό το γνωστό φυτοφάρμακο και από αυτές τις έξι μελέτες ορισμένες ε, δεν δημοσιοποιήθηκαν καν και εγώ εδώ αναρωτιέμαι είναι σοβαρά τα επιστημονικά αυτά δεδομένα μάλλον όχι ε, τα επιστημονικά δεδομένα στα οποία βασίζει το σχέδιό της Κομισιόν για να επιτρέψει για άλλη μια δεκαπενταετία αυτή τη χημική ένωση. Η, άποψη της ΕΦΣΑ ε, συνάδει με τα όσα υποστήριξε και η ΆΡΚΑ η οποία έκανε μια σοβαρή επιστημονική μελέτη η οποία καταδεικνύει ότι αυτή η χημική σύνθεση δημιουργεί βλάβες στο DNA και στα χρωμοσώματα σε ανθρώπινα κύτταρα. Οπότε θα ήθελα εγώ η άποψη της Κομισιόν, το τελικό κείμενο, να λάβει υπόψη όχι μόνο την άποψη της ΕΦΣΑ, την οποία θεωρώ ανεπαρκώς επιστημονική, αφού απλά κάνει μια αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων, δεν ε, βασίζεται σε σοβαρές ε, επιστημονικές μελέτες. Οπότε θα ήθελα να ακολουθήσετε αυτή την οδό για την προστασία της υγείας των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα 5.000 γεωργοί ε, διαμαρτύρονταν στο Ελσίνκι λόγω της κατάστασης στην γεωργία. Όπως γνωρίζετε, η Φιλανδία έχει μακρά παράδοση εμπορικών συναλλαγών με την Ρωσία και ιδιαίτερα όσον αφορά τα γαλακτοκαμικά προϊόντα. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι η Γενική Διεύθυνση Σάντε τι κάνει για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εξάγουν τρόφιμα προς την Ρωσία προϊόντα που δεν βρίσκονται στον ε, κατάλογο ε, του εμπάρκου. Για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά χωρίς λακτόζη. Επίσης, υπάρχει η διαμάχη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας ASF. Ε, τι γίνεται λοιπόν όσον αφορά τα προϊόντα χειρίου κρέατος σε σχέση με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Δύο ζητημάτα. Πρώτον, κανείς δεν ανέφερε την υγεία και την ευημερία των αγροτών και των οικογενειών τους. Ξέρετε, εμένα με απασχολεί παρότι δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα, η ευημερία των αγροτών μας, αλλά και το επίπεδο των ατυχημάτων, τραυματισμών και θανάτων που υφίστανται οι αγρότες για να παράγουν τα φαγητό που τρώμε. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη και αυτό το ζήτημα και θα έχετε τη δική μου υποστήριξη. Το δεύτερο αφορά το αλογισιο κρέα. Υπάρχει μια περίεργη κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει αλογισιο κρέα από το Μεξικό και τον Καναδά και παρακολουθεί το κρέας αυτό μόνο έξι μήνες πριν αυτό εισαχθεί. Ωστόσο, τα κρέατα, τα αντίστοιχα των αλόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται ε, ε, ε, πιο αυστηρές απαιτήσει. Πολλά αλόγα δεν μπορούν να μπουν στην διατροφική αλυσίδα παρότι θα μπορούσαν. Οπότε έχουμε σπαταλή μόνο έτσι, μπορεί να έχουμε και ζήτημα καλής μεταχείρισης των αλόγων. Έχετε κάποια λύση, γνωρίζετε το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, εξαντλήσαμε το κατάλογο των ομιλητών. Α, και ο κύριος Εκ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Εκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των κουνελιών, αλλά νομίζω ότι αυτό το καλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Άλλη ερώτηση λοιπόν. Πρόκειται για θέμα υγείας και των ανθρώπων. Έχετε σκεφτεί σε τι βαθμό βλάπτεται η ανθρώπινη υγεία από τους φίλους των ζώων με αυτά που συμβαίνουν στον γεωργικό τομέα. Ε, ένα κοριτσάκι την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε σχεδόν κλαίγοντας στην πόρτα μου. Ε, το διαδίκτυο ε, είναι ευλογία, είναι όμως και κατάρα, διότι όλες οι παραβιάσεις που πραγματοποιούνται μέσα σε τρεις-τέσσερις ώρες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν ε, πάνε σε γιατρούς ε, λόγω αυτών που βλέπουν στο διαδίκτυο και αυτά ε, συνδέονται με τον τομέα εργασία τους, σε την δημόσια υγεία. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να το σκεφτεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν θέλετε το λόγο. Γιατί θέλω να εξηλωθώ για την πρωινή μας ε, μικρή διαμάχη. Δεν θέλετε. Οκ, okay, εντάξει. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος ε, Αντριουκάητο, ο Επίτροπος, έχει το λόγο για να απαντήσει. Okay, may I start with... Ωραία. Να ξεκινήσω από την ερώτηση της κυρίας Σταμάτο για την ξύλα λαφαστιδιόζα. Και ο κύριος Καπούτο έθεσε το θέμα αυτό. Θέλουμε επιστημονικά επιχειρήματα. Έχουμε τα επιχειρήματα της ΕΦΣΑ. Είναι απόλυτα σαφής η κατάσταση. Θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσετε τις σχετικές νομοδοτήσεις να τις συζητήσετε μεταξύ σας. Διότι μόνο έναν επιστημονικό φορέα έχουμε στην νομοθεσία μας. Είμαι υποχρεωμένος να ακολουθώ την νομοθεσία και να ακολουθώ τις διαδικασίες που σχετίζονται με το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί και από τις δύο πλευρές, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Διότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δημιούργησαν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Πιο, σχετικά δηλαδή με το ποιος είναι αρμόδιος για τις επιστημονικές νομοδοτήσεις και για τις επιστημονικές αξιολογήσεις. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις για τα φυτοφάρμακα, η ΕΦΣΑ είναι αρμόδια. Όσον αφορά λοιπόν την ξυλέλα, ακολουθούμε τα επιστημονικά στοιχεία. Και πάντα ζητούμε από την ΕΦΣΑ να εξετάσει τα νέα επιστημονικά στοιχεία και να τα επικαιροποιεί, να επικαιροποιεί τις νομοθετήσεις της με βάση τα νέα στοιχεία. Εάν λοιπόν έχετε νέα στοιχεία να μας τα στείλετε, να τα στείλουμε στην ΕΦΣΑ για να τα ε, αξιολογήσει. Εγώ λοιπόν ε, έχω την υποχρέωση να ακολουθώ τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Συνέχεια μου λέτε ότι δεν πιστεύετε την ΕΦΣΑ. Τότε θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία μας. Να προτείνετε κάτι καινούριο. Αυτό όμως είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τι θέλετε λοιπόν να κάνω, διότι πρέπει να ακολουθούμε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ομοθεσία και που βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Εγώ, με την ιδιότητά μου, δεν μπορώ να παραβιάσω τον νόμο. Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε τα διάφορα μέτρα. Έχουν γίνει έλεγχοι της Επιτροπής στην Ιταλία και στην Γαλλία για να εξετάσουμε ε, την εφαρμογή των επιγόντων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει νομική διαμάχη ε, την Πούλια, στην Ιταλία σχετικά με εγκληματικές ενέργειες. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να ακολουθούμε αυστηρά τις δικές μας διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση με βάση τα επιστημονικά στοιχεία. Είμαι διατεθειμένος ε, να συζητήσω μαζί σας ε, όλα τα θέματα αυτά ε, αναλυτικά. Όσον αφορά την επισήμανση του μελιού. Γνωρίζετε ότι είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Δεν είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας, αλλά ευχαρίστως να μεταφέρουμε τις θέσεις σας όσον αφορά την επισήμανση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς ε, για την κατάσταση στον τομέα του μελιού. Όσον αφορά τον αμίαντο, ε, εργαζόμαστε πολύ στενά με τον ε, αρμόδιο επίτροπο και Είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε το θέμα εις βάθος. Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, θα μεταφέρω τι θέσει σα ε, στον Επίτροπο Δέλα. Είναι όμως η υποχρέωσή μας να συνεργαζόμαστε, διότι το θέμα του του συνδέεται στενά με τα θέματα περιβάλλοντος. Όσον αφορά την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, θα ήθελα να σας πω το εξής όταν μιλάμε για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν οργανώνουμε συνεχώς σε συναντήσεις, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά σε υψηλό επίπεδο. Στο Βίλνιους είχαμε πρόσφατα σχετική συνάντηση, όπου οι επακεφαλής των κτηνιατρικών υπηρεσιών ε, τεσσάρων χωρών ε, παραβρέθηκαν και συζητήθηκαν και οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και άλλη συνάντηση ε, στο Ταλίν ε, με την Λετωνική, Λιθουανική, ε, με τους υπουργούς Λιθουανίας, Εστονίας και Λετωνίας και Πολωνίας. Επίσης η Φιλανδία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία έστειλαν εμπειρογνώμονες. Έχουμε προβλήματα στα σύνορα και γι' αυτό θέλουμε να προειδοποιήσουμε τις χώρες που δεν έχουν ακόμα προβλήματα στον τομέα αυτών ότι είναι σημαντικό να αρχίσουν να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα για το θέμα αυτό. Αναφερθήκατε σε οικονομικά μέσα. Νομίζω ότι αυτά εμπίπτουν στην κοινή γεωργική πολιτική, άρα αρμόδιος είναι ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν. Όσον αφορά όμως τα ευέλικτα μέτρα και την εφαρμογή τους για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανόλης των χείρων σε περιοχές που έχουν πληγεί από αυτήν την ασθένεια, βασίζουμε τις ενέργειές μας σε συγκεκριμένες Έρευνε που πραγματοποιούνται κάθε μήνα. Όσον αφορά τις ζώνες 2 και 3, προσπαθούμε να ανακουφίσουμε τις εκμεταλλεύσεις με την εφόσον εφαρμόζουν τα μέτρα. Το φθινόπωρο σκοπεύουμε να οργανώσουμε μια σημαντική συνάντηση στην Πολωνία. Η Πολωνία δέχθηκε να οργανώσει τη συνάντηση αυτή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας να βοηθούμε τους γεωργούς και τις ε, μεγάλες εκμεταλλεύσεις για την επίλυση του προβλήματος. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι ο έλεγχος του πληθυσμού αγριόχειρων. Αυτό είναι το θέμα που θα πρέπει να μας αποσχολήσει και είμαστε διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Πάντως, ε, Έχουμε διαδικασία για την διαχείριση της κατάστασης. Επίσης, ε, στον κύριο Γιάρ να απαντήσω για τη γλυφοσάτη, το ρωσικό εμπάρκο και τον μαύρο κατάλογο Ρώσων Υπουργών. Είχα συναντήσεις με την αντιπροσωπεία της Ρωσίας εδώ στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε τη δυνατότητα διοργάνωσης μιας κοινή συνάντησης και για να συζητήσουμε περισσότερο ει βάθο τα θέματα αυτά. Από την άλλη μεριά έχουμε τη διαμάχη στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Το θέμα αυτό βρίσκεται στα χέρια μας και πρόκειται να το προωθήσουμε. Και αναφερθήκατε και στο θέμα της γλυφοσάτης ε, και της αποχής ε, κάποιων κρατών μελών. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, και πάλι στο εξής. Τα κράτη-μέλη στη Μόνιμη Επιτροπή υποβάλλουν τις θέσεις τους και είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να την συζητήσουμε. Όπως γνωρίζετε, οι κάτω χώρες πρότειναν να εισαχθούν κάποια προσωρινά μέτρα, να έχουμε έρευνες ε, του Οργανισμού Χημικών του Χρόνου. Κάποια κράτη-μέλη διαφωνούν, να είμαστε διατεθειμένοι όμως να το συζητήσουμε αυτό με τα κράτη-μέλη, καθότι έχουμε χρόνο και με βάση την αρχή της προφύλαξης είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα θα ήθελα να επαναλάβω επειδή το επισήμαναν πολλοί ευρωβουλευτές το ότι η νομοθεσία που έχουμε και που κατοχυρώνεται και στις εθνικές νομοθετικές τάξεις προβλέπει ότι η βιομηχανία έχει δικαίωμα να υποβάλει μελέτες καλύπτονται από την ρήτρα του απορρίτου, της εμπιστευτικότητας. Εγώ πρότεινα στη βιομηχανία να δημοσιεύσουν αυτές τις μελέτες και ελπίζω να δεχτούν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας το αίτημα να δημοσιεύσουν αυτές τις μελέτες. Πάντως προστατεύονται από τη ρήτρα της εμπιστευτικότητας που κατοχυρώνεται στο νομοθετικό μας πλαίσιο. Βέβαια, μπορούμε να τροποποιήσουμε την νομοθεσία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα και να ζητούμε από τη βιομηχανία δημοσίευση τέτοιων μελετών. Γιατί καλό θα ήταν να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο κύριος Αντριέ αναφέρθηκε στο θέμα της γρήπης των πουλερικών. Το συζητήσαμε αυτό το πρόβλημα και με τον Γάλλο Υπουργό. Αφορά πάπιες και χήνες. Είναι διαφορετική η γρήπη των πουλερικών στις πάπιες και τις χήνες από ό,τι στα πουλερικά. Γιατί οι πάπιες και χήνες δεν έχουν συμπτώματα λίμωξη, μόλυνσης. Πάντως το θέμα είναι ευρύτερο και θα πρέπει να συνεργαστούμε για να σημειώσουμε πρόοδο. Πάντως οι γαλλικές αρχές ε, έχουν αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την γρήπη των πουλερικών ε, είναι πολύ αξιόλογο και πιστεύω ότι η Γαλλία θα καταφέρει να ξεριζώσει αυτή τη ζωονόσο στις πληγήσεις περιοχές. Πάντως, ο Υπουργό θα ξαναεπισκεφτεί αυτές τις περιοχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πραγματοποιήσει τέτοια επίσκεψη για να βοηθήσουμε τη Γαλλία να εξαλείψει αυτή τη ζωονόσο τη γρήπη των πουλερικών, κυρίως στις πάπιε και χήνες. Αναφέρθηκε και το ερώτημα του ευνοχισμού των χείρων και το θέμα του αίματος από φοράδες και τη χρησιμοποίηση του στη χειροτροφία. το αίμα ε, έγκυων φοράδων που χρησιμοποιείται στη χειροτροφία. Ε, επισημάνθηκε πιθανή κακή μεταχείριση των φοράδων, κυρίως σε τρίτες χώρες. Πάντως, οι κανόνε του ΠΟΕ προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει τις δικέ προδιαγραφές καλής μεταχείρισης των ζώων στι τρίτες χώρες. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους για να έχουμε κοινή αντίληψη των προδιαγραφών της καλής μεταχείρισης σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό ενδεχομένω θα αναβαθμίσει τι προδιαγραφέ καλή μεταχείρισης γενικώ. Πάντως ε, έχουμε ε, ε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων έχει ε, αντίστοιχα καλές προδιαγραφές και η χρήση ε, των ζώων για ερευνητικού σκοπούς καλύπτεται. Είναι έτοιμος και ο φορέας αυτός να παρακολουθεί την κατάσταση και να ενθαρρύνει τις διάφορες χώρες να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές του ΠΟΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ευνοχισμό των κάπρων. Υπάρχει δυνατότητα για χειρίδια ε, κάτω των 7 ημερών να υπόκειται σε ευνοχισμό χωρίς αναισθησία. Εξετάζουμε αυτό το θέμα της ε, χορήγης παυσιπώνων ή αναισθητικού σε όλα τα χειρίδια. Περιμένουμε τα πορίσματα αυτές τις μελέτες το Φεβρουάριο του 2017 και στο μεταξύ θα προωθήσουμε ε, τρόπους για ανώδυνο ευνοχισμό των χειριδίων. Κάποιοι ευρωβουλευτές ανέφεραν το παράσιτο μαύρη κοιλίδα στα εσπεριδοειδή, το black spot. Τα κράτη-μέλη έλαβαν ε, κάποια μέτρα κατά της Νοτιοαφρικής και κατάφεραν να μην εισχωρήσει η μαύρη κοιλίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είχαμε επίπονες συζητήσεις με την Νοτιοαφρική και τον Διεθνή Οργανισμό για την Προστασία των Φυτών. Συνεχίζεται η συζήτηση για το πώς θα συνεχίσουμε τις πιέσεις προς τη Νότια Αφρική για να επιληθεί του ζητήματος της εξάλληψης ε, της μαύρης κοιλίδας ε, στα εσπεριδοειδή. Τώρα, για την κατάσταση στη Ρουμανία. Έχουμε καλή συνεργασία με τη Ρουμανία και υπάρχει πρόοδος. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διμέρειες συζητήσεις. Ε, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για πρόοδο. Η κυρία ε, Γκαρσία, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε έγγραφο εργασίας με αυτό το αντικείμενο, με τα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ε, εφαρμόζουμε τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και μετά και τον οδικό μας χάρτη θα οργανώσουμε καλύτερα τις συζητήσεις με τους εμπειρογνώμονες και μάλιστα και αναμένεται για τον επόμενο μήνα ένα σχέδιο θέσεις ε, για τα κριτήρια των εδοκρινικών διαταρακτών ακολουθώντας τους ορισμούς ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Η κυρία Μαγκίνες αναφέρθηκε στην υγεία και ψυχική υγεία των αγροτών. Όπως ξέρετε, έχουμε πλατφόρμες για την ψυχική υγεία και αρχίσαμε και ασχολούμαστε και με αυτό το θέμα. Και στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ προσπαθούμε να βρούμε πιο συγκεκριμένους τρόπους ε, για να λάβουμε υπόψη τις ειδικέ ανάγκες, ε, κυρίως των ηλικιωμένων, στην Ήπεθρο. Αναφερθήκατε και στο αλογίσιο κρέας από το Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, έχουμε επίγνωση του προβλήματος, ε, έχουμε και συνεδριάσεις σχετικές και μάλιστα υπάρχει μια διαφορά με το Μεξικό αυτή τη στιγμή γιατί θεσπίσαμε περιοριστικά μέτρα κατά των εισαγωγών αλογίσιου κρέατος από το Μεξικό. Και παρακολουθούμε την κατάσταση επί τόπου. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με τον Καναδά και τη μεταφορά λόγων από τις Ηνωμένε Πολιτείες στον Καναδά και μετά την εξαγωγή του αντίστοιχου κρέατος και αυτό το θέμα το εξετάζουμε επισταμένος. Πάντως ως προς το Μεξικό έχουμε απαγόρευση των εισαγωγών αλογίσιο κρέατος από το Μεξικό. Η κυρία Χάζακα ανέφερε ζητήματα περιστρατηγικών ε, για την καλή μεταχείριση των ζώων και πρέπει να πω ότι έχουν γίνει αναλυτικές ε, διεξοδικές συζητήσεις στο Συμβουλίο Γεωργίας και είναι τόσο πολλές και διαφορετικές οι απόψεις των κρατών μελών σε σχέση με την εισαγωγή, για παράδειγμα, νέων νομοθετικών προσεγγίσεων είναι ε, οι προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε για μια νέα στρατηγική ε, καλής μεταχείρισης των ζώων. Αυτή τη στιγμή ε, ετοιμαζόμαστε, ετοιμάζεται να δημοσιευθεί η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου και μετά θα υλοποιήσουμε όλα τα μέτρα που σχετίζονται με, τις παλιότερες, με την παλιότερη στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων. Οκτώ μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί και έχουμε έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες κινήσεις ώστε να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μέχρι το 2017 αλλά ξέρετε και έχουμε και ένα διάλογο με τους ενδιαφερομένους αλλά κατά την απόψή μου πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα για την καλή μεταχείριση των ζώων. Θα είναι ένας οργανισμός που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και θα συζητήσει και την πορεία που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον ε, σε σχέση με μια νέα στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων. Τώρα, όσον αφορά αυτή την πλατφόρμα, και εκεί ε, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει άλλη άποψη. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή άποψη. Αλλά εμεί θέλουμε να καλέσουμε τα κράτη μέλη εκείνα τα οποία δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την πλατφόρμα ε, τη καλή μεταχείριση των ζώων. Ε, να καλέσουμε λοιπόν αυτά τα κράτη μέλη να ιδρύσουν αυτή την πλατφόρμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να διευκολύνει, να βοηθήσει στην ε, δημιουργία τη. Συγγνώμη, αλλά περνάει ο χρόνο και Τώρα, να απαντήσω μια ερώτηση σε σχέση με τους γεννατικά τροποποιημένους οργανισμούς. Για άλλη μια φορά η Επιτροπή λυπάται που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την νομοθετική της πρόταση. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο. Η πρότασή μας ήταν η ίδια με τα ζητήματα των καλλιεργιών. Τα ίδια ακριβώς προτείναμε για τις γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για τρόφιμα και ζωοτροφές. Και όπως γνωρίζετε τώρα, το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συζητήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Εξετάζουμε εμείς τις θέσεις του Συμβουλίου. Η συζήτηση πιστεύω θα πρέπει να συνεχιστεί πιο επικοδομητικά. Και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε κάποιες βελτιώσεις στην τρέχουσα κατάσταση, η οποία μοιάζει με έναν ε, ε, διάλογο καταδικασμένο στην αποτυχία. Διάλογο κουφών. Ε, ε, το Κοινοβούλιο ε, απέρριψε την πρότασή μας. απέριψε την πρότασή μας να αναλάβουμε ευθύνη σε επίπεδο κρατών μελών επίσης. Να αναλυθεί ευθύνη και από τα κράτη-μέλη επίσης. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσετε την ευκαιρία για αυτή την εμβριθή ανάλυση που ήταν και αρκετά χρονοβόρα. Αλλά τα πιο δύσκολα θέματα τα αφήσαμε για το τέλος. Τα τόσο ευχάριστα θέματα που απασχολούν τόσο πολύ τους συμπολίτε μας. Πάντως σας ευχαριστώ θερμά γιατί ήταν ευρυθής και πολύ σοβαρή και σημαντική αυτή η συζήτηση και σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έχουμε πολύ, δύο πολύ σημαντικά θέματα, την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου, το επόμενο μας θέμα, και τις διαπραγματεύσεις στο TTIP. Πολύ σημαντικό θέμα γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε τις προδιαγραφές μας για τα τρόφιμα. Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά κύριε Επίτροπε. Ε, ευχαριστούμε και το συνεργάτη σας. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο της ημέρησης διάταξης. Νομίζω ότι εκπληρώσαμε τις απαιτήσεις του διαρθρωμένου διαλόγου και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Επίτροπε. Είστε έτοιμοι, έτοιμος κύριε Γιάρ για το επόμενο θέμα. τύμπερ της μετακλογικής αναθεώρησης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί θέλουμε να προλάβουμε την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ετοιμάσουμε τη δική μας θέση για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Δύο είναι οι αρμόδιοι ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Προπολογισμών ο κύριος Όλμπρεχτ και η κυρία Τομά, Τωμά. Και από εμά θα συντάξει γνωμοδότηση ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συζητήσεις, γιατί θα πρέπει να δώσουμε και το δικό μας στίγμα, τις δικές μας προσδοκίες, τις δικές μας απόψεις ε, για την ενδιάμεση αναθεώρηση και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα κοφεύσει απέναντι στα αιτήματά μας και στις παρατηρήσεις μας. Και καλό είναι να έχουμε ελπίδα και να είμαστε αισιόδοξοι. Κύριε Γιάννη, έχετε το λόγο. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα θα αναφερθώ στο θέμα διότι μας πιέζει ο χρόνος. Ελπίζω ότι αργότερα θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο εκτενή συζήτηση. Πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας. Μιλάμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στους συναδέλφους να πω διότι με ρώτησαν αρκετοί ποιο είναι το νόημα αφού έχουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, το νέο είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων, πρέπει λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε ε, κατόπιν συνεννόησης με τους συναδέρφους μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμούς. θα ήθελα να προτείνω τα εξής. Πρώτον, να είναι σχετικά σύντομη η γνωμοδότηση. Αυτή στόχο είναι να παραμείνουμε εντό των 10 σελίδων, ε, καλύτερα να, πούμε συγκεκριμένα τι θέλουμε και να παραμείνουμε εντό θέματος. Ε, η πρώτη μου επιθυμία λοιπόν θα ήταν να έχουμε μια κοινή θέση και η δεύτερη επιθυμία μου είναι να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές ε, εμείς από το τομέα της γεωργίας. Πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα λοιπόν να ζητούμε πόρους για αυτά που ζητάει από μας η κοινωνία. Εάν η κοινωνία ζητάει περισσότερα από εμά, χρειαζόμαστε και περισσότερα χρήματα για να τα εφαρμόσουμε. Και θα πρέπει να προβλέψουμε νέα αποθεματικά λόγω της αστάθειας των τιμών διότι τα ε, ισχύοντα μέσα ε, για τη σταθερότητα δεν αρκούν. Η πρότασή μου όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα είναι η εξή. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. 6 Ιουνίου ε, η ψηφοφορία στην άκρη. Ήδη σήμερα ε, έχουμε την προθεσμία της τροπολογίας 29 Απριλίου. Μέχρι τότε μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Εγώ θα πρότεινα ήδη στις 22 Μαρτίου να έχουμε μια πρώτη συνάντηση σκιωδών εισηγητών. Θα παρακαλούσα την ε, γραμματεία να μου δώσει τα ονόματα των σχεδόν εισηγητών από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Να έχουμε λοιπόν μια πρώτη στρατηγική συζήτηση και μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθω σε επαφή με τους ε, συναδέλφους, τους κοιόδες εισηγητές, θα τους στείλω ένα πρώτο σχέδιο κειμένου και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε για να εκπονήσουμε τη γνωμοδότηση. Στόχος μας ε, θα είναι στο τέλος γνωρίζοντας και όλους ε, τους συναδέλφους μας ε, να έχουμε μια γνωμοδότηση με ευρία υποστήριξη και με αυτή να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμού η ευρεία πλειοψηφία θα μας δώσει και την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Αυτά εισαγωγικά. Ίσως θα μπορέσουμε αργότερα να έχουμε και συζήτηση επί του περιεχομένου. Θα στείλω λοιπόν το έγγραφό μου στους σκιώδεις εισηγητές. Συνοψίζω λοιπόν να παραμείνουμε εντό θέματος, το μήνυμά μας σε λίγες σελίδες να το μεταφέρουμε και να έχουμε ευρία υποστήριξη ώστε να μπορέσουμε με αυτοπεποίθηση να διαπραγματευτούμε. Έχουμε επιδείξει δημοσιονομική πειθαρχία, ε, ήμασταν συνεπείς στη θέση μας. Ε, ελπίζουμε λοιπόν ε, οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Προϋπολογισμού να μας ανταμείψουν γι' αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ ξεκίνησε τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους ε, εισηγητές. Θα συνεχιστούν φυσικά. Οπότε σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση, αλλά μην διστάσετε να στείλετε και τις προτάσεις στον κύριο Γιάρ. ώστε να συγκεντρώσει το υλικό από την Επιτροπή μας για να προσδιορίσουμε τις δικές μας προσδοκίες για την κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο. Δεν βλέπω ακόμη κανέναν εθελοντή. Περιμένω. Η ε, κυρία Πετήρ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάρ για την προσέγγιση του που πήρε πολύ στα σοβαρά το έργο του και θα λάβει υπόψη τα δικά μας ενδιαφέροντα και τις προτάσεις και το συμφέρον φυσικά των γεωργών μας. Εγώ πρώτη φορά ε, βλέπω τέτοια προθυμία και χαίρομαι ιδιαίτερος. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ο κύριος Γιάρ να κρατήσει τη γραμμή της ε, διατήρησης του γεωργικού προϋπολογισμού, να μην γίνουν περαιτέρω περικοπές. Θα ήταν πολύ αρνητικό να διαταραχθεί ο γεωρικός προϋπολογισμός και ενθαρρύνω τον κύριο Γιάρ ε, να τονίσει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οικογενειακές, ε, οι μικρές εκμεταλλεύσεις για τη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας, τη προστασία του περιβάλλοντος, για την παραγωγή των τροφίμων, αλλά και για τη διατήρηση των παραδόσεων στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον. <coughs> Ναι, κύριε Πρόεδρε, αυτό δείχνει την αυτοπεποίθηση της Επιτροπής, πόση εμπιστοσύνη έχει στον κύριο Γιάρ ε, η Επιτροπή. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ ικανός ικανό μέλος του Κοινοβουλίου αυτού και ξέρουμε ότι θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι τεράστια ευθύνη και υπάρχουν ε, πολλές δυσκολίες τώρα στα γεωργικά ζητήματα και είναι δύσκολο να μιλά κανείς για προπολογισμού όταν ο κόσμο πονάει αλλά του έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα επιτελέσει εξαιρετικό έργο και είπε πολύ σωστά ότι οι σκιώδεις ε, θα πρέπει να συνεργαστούν πολύ στενά μαζί του ε, για να γίνει εξαιρετική δουλειά εκ μέρους της Επιτροπής και ε, για λογαριασμό της ε, γεωργίας των γεωργών. Θα δούμε τι θα μου πείτε όταν θα υποβάλει το έγγραφό του ο κύριος Γιάρ. Τότε να δείτε ε, πόσες τροπολογίες ε, θα υποβληθούν και εκεί θα κρίνουμε πόσο συμφωνείτε με την προσέγγιση του κυρίου Γιάρ. Η κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιάρ, εγώ θα είμαι σκιώδη από την ομάδα μου και ελπίζω να συμβάλλω στην εκπόνηση μιας καλής έκθεσης. Δεν είχα ζητήσει στην αρχή το λόγο γιατί δεν κατάλαβα ότι θα γινόταν συζήτηση. Γιατί νόμιζα ότι δεν θα γινόταν σήμερα η συζήτηση. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε μη τι άλλο το γεωργικό προπολογισμό στο σημερινό επίπεδο. Αυτό είναι ο πρωταρχικό μα στόχο. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τον προπολογισμό τη γεωργία, να μην υποστεί άλλε περικοπέ. Και αυτή είναι η βασική δυσκολία ίσως που θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί όπως φαίνεται στο Συμβούλιο δημιουργήθηκε εντύπωση και αυτό διαβάσαμε στον τύπο ότι υιοθετήθηκαν νέα μέτρα και θα υποβληθούν νέα μέτρα ε, για τη Γεωργία. Ε, νέα μέτρα για τη Γεωργία. Αλλά τίποτα δεν αναφέρθηκε για τη χρηματοδότησή του. Δεν υπάρχουν, νέα, δεν προβλέφθηκαν νέα κονδύλια. Δεν μπορούμε χωρί νέα κονδύλια να αντιμετωπίσουμε και τι συγκυριακέ και τι διαρθρωτικέ ανάγκε τη γεωργία. Συμφωνώ να είστε ε, συνοπτικός στο έγγραφό σα, να επικεντρωθείτε στα ουσιώδη, ούκεν το πόλο το εφ, και να είναι και πιο ισχυρή η φωνή μας. 22 Μαρτίου θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση, συνάντηση εργασίας, αν δεν κάνω λάθος μαζί σας. Έτσι κύριε Γιάρ, μάλιστα. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον συνάδελφο, στον κύριο Γιάρ και πιστεύω ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έγγραφο αυτό να έχει τη σωστή προοπτική. Η κατάσταση στη Γεωργία είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε για αναθεώρηση και διόρθωση, ε, δεν είναι κάτι αμεληταίο. Όλοι λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν ευθύνεται η Γεωργία για την κρίση, ούτε για τα προβλήματα των εξαγωγών ε, ε, στη Ρωσία. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στη διπλωματία. Σε προβλήματα διπλωματίας. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να πληρώσει την ύφη η Γεωργία ούτε να γίνει από τράχος λόγω αυτών των προβλημάτων. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναζωογονήσουμε τα αγροκτήματα. Έχουμε περιορισμένο ε, χρηματικά ποσά. Ε, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες πιστώσεις ή κάποια ε, συστήματα εγγυήσεων, να ψάξουμε να βρούμε κάποιες επιπλέον λύσεις, ώστε οι γεωργοί μας να πιστέψουν ότι θα είναι επωφελής αυτή η αναθεώρηση για αυτούς. Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη και προσβλέπουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να περάσουμε στο τελευταίο σημείο για να, σχετικά γρήγορα για να έχουμε περισσότερο χρόνο στη συζήτηση. Ο κύριος Άγνιο. Right, well, uh, λοιπόν, για να ταράξω λίγο τα νερά εδώ όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020 σε 100 ημέρες το Ενωμένο Βασιλείο θα ψηφίσει αν θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη τη στιγμή θα χρειαστεί να δείτε τι θα κάνετε χωρίς τη δική μας συμβολή μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ε, απλά το επισημαίνω γιατί θα αποτελέσει πονοκέφαλο για όλους ε, ελπίζετε βέβαια ότι θα μείνει ε. ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε αλλά από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Ερντός, καταλάβουμε ότι ήδη έτσι είναι η κατάσταση, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα. Ο κύριος Ντές, παρακαλώ, χρόνο φίδου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Χαίρομαι που ο κύριος Γιάρ έχει αναλάβει το θέμα αυτό και ε, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν και θα τον στηρίξουμε όσο μπορούμε. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση όσον αφορά τα κονδύλια για την γεωργία. Όλο τίθεται το θέμα γιατί η Γεωργία λαμβάνει το 40% των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αν είχαμε αναλογική κατανομή, τότε η Γεωργία θα, θα λάμβανε το 1%. Αλλά για τον ε, τομέα που παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα του τα τρόφιμα, αυτό θα ήταν πάρα πολύ λίγο. Θέλουμε να διατηρηθεί η παρούσα χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνη είναι και η τελευταία. Για το θέμα των 100 ημερών. Είναι απόφαση των, Ευρωπα... των Βρετανών πολιτών. Πάντως την εκατοστή πρώτη μέρα ούτω ή άλλω τα κονδύλια θα εισρέψουν γιατί ακόμη και αν ε, αποφασιστεί αποχώρηση θα χρειαστεί κάποια διαδικασία γι' αυτό. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χέισλερ, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά παρακαλώ να είστε λακωνικός. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη διαδικασία. Έχουμε την διοργανική ε, συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση, την ε, εκπονούμε αυτή τη στιγμή και ε, έχουμε προθεσμία για την ολοκλήρωσή της μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το Κοινοβούλιο ζήτησε στην ενδιάμεση αυτή ε, αναθεώρηση να εξεταστούν πιθανές νέες πρωτοβουλίες και να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει συζήτηση σχετικά με το αν χρησιμοποιούνται με σκόπιμο και στοχευμένο τρόπο οι πόροι. Υπάρχει σημαντικός περιορισμός για τον τομέα της γεωργίας. Γνωρίζετε ότι εσείς μαζί με το Συμβούλιο αποφασίσατε η κατανομή στα κράτη-μέλη ε, στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής να μην αποτελέσει αντικείμενο αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης. Μπορώ λοιπόν να στείλω καθησυχαστικό μήνυμα στον τομέα της γεωργίας. Το θέμα δεν θα είναι ε, αν θα δοθούν περισσότερα ή λιγότερα χρήματα στη γεωργία. Δεν θα θυχθούν οι πόροι της γεωργίας. Επίσης, στη συζήτηση ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο να συμπεριλαμβάνονται περισσότερα στην έκθεση αυτή ε, σχετικά με τα αποτελέσματα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης, επιτέθησαν οι στόχοι, ε, και στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής ε, θα γίνει η σχετική συζήτηση. Ο η συγητής Όλπριχτ έχει θίξει το θέμα και νομίζω θα είναι κεντρικό θέμα στην πολιτική συζήτηση. Γνωρίζετε ότι η σημαντική προτεραιότητα του Επιτρόπου Χόγκαν είναι η απλοποίηση στην διάμεση αυτή έκθεση. Στον βαθμό που είναι δυνατόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιφέρουμε απλοποιήσεις στην κοινή γεωργική πολιτική μαζί με άλλες πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες από την εφαρμογή της πολιτικής. Στον τομέα της γεωργίας ε, νομίζω ότι διαγράφεται μία προτεραιότητα. Ακριβώς αυτή η απλοποίηση. Όσον αφορά το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης όσον αφορά τις ε, νέες δημοσιονομικές προβλέψεις. Η Κομισιόν θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2017 να υποβάλει σχετική πρόταση. Οι συζητήσεις λοιπόν θα διεξαχθούν ε, κατά τη διάρκεια του έτους. Και θα έχουμε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής και το μέλλον της χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν είναι επί του παρόντος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ένα λεπτό κύριε Γιάρδο, δεν νομίζω ότι έχει, υπάρχει ανάγκη για πιο εκτεταμένη δευτερολογία. Ναι, να σας ευχαριστώ καταρχάς για την εμπιστοσύνη σας όσον αφορά την εκπόνηση της έκθεσης αυτής και στην Επιτροπή Γεωργίας. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με ευρία πλειοψηφία να υιοθετήσουμε την έκθεση. Προσβλέπω στην πρώτη συνάντηση των σκηνησυγητών στις 22 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Μέχρι το τέλη Απριλίου έχετε διορία για την υποβολή τροπολογιών. Περάμε στο επόμενο θέμα, τις διαπραγματεύσεις του TTIP που προβλέπονται η σχετική συζήτηση να γίνει και κλεισμένων των θυρών. Η γραμματεία θα μου πει ποιοι δικαιούνται να παραμείνουν στην αίθουσα σε μια και κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.